Okay, good evening, colleagues. Um, Καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εφόσον δεν έχετε ε, αντιρρήσεις, η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Τώρα, δεν έχουμε διερμηνία στα κροατικά, τα μαλτέζικα, τα δανέζικα, τα ιρλανδέζικα και διάφορες άλλες γλώσσες, αλλά στα ελληνικά υπάρχει. έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης 21-22 Δεκεμβρίου 20, ε, του 2015 και 19 Μαΐου 2016. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα και αν δεν υπάρξει αντίρρηση από πλευρά σας θα εγκριθούν. Καθίσατε να ξεκινήσουμε. Έχετε ένα διαδικαστικό, κύριε Άλβιο. Ναι, παρακαλώ. Δεν έχω την ε, κάρτα μου, τη φέρνουν. Μπορώ στο ξεκίνημα τόσο να ψηφίζω διανατάσεως της χειρός. Θα προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία, οπότε να σηκώνετε το χέρι σας. Αυτό αρκεί. Θα ήθελα να τσεκάρω αν έχετε όλοι οι υπόλοιποι την κάρτα ψηφοφορία σα. Είναι κανεί που δεν την έχει μαζί του. Ωραία. Προχωρούμε. Με εξαίρεση την κυρία Άλπιο που θα σηκώνει το χέρι της. Σημείο 4. Ευρωπαϊκή συνοριακή, ε, ε, συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Έκθεση Πάμπρεξα. Η προσωρινή συμφωνία για το φάκελο αυτό, συνάδελφοι, επιτεύχθηκε στο ημερή διάλογο στις 21 Ιουνίου. Σήμερα ψηφίζουμε για την, έκβαση, για την έγκριση της έκβασης των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 73.5 του κανονισμού. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή εντάχει για ένα σύντομο σχόλιο και κατόπιν θα προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Κύριε Πάμπρεξ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους κοιόδης συζητητές. Είχαμε κάνει μια πολύ επικοδομητική δουλειά. Τελειώσαμε το... την έκθεση σε τέσσερις μήνες. Το έγγραφο αυτό επιτρέπει τη δημιουργία μιας υπηρεσίας που θα αλλάξει την κατάσταση. Και δεν το λέω πολιτικά, το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ασφαλέστερη Ευρωπαϊκή Ένωση με καλύτερη διαχείριση των συνόρων μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αν κάποιοι αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να τους παραπέμψετε στους και ηγητές μας ε, που διαπραγματεύτηκαν αυτοί, αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ κύριε Πάμπριξ θα περάσει, εάν εγκριθεί το κείμενο θα περάσει στην ε, Ολομέλεια, στην ε, επόμενη, σε επόμενη σύνοδο. Θα κάνουμε μία ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κείμενο του τριμερούς διαλόγου βάσει του άρθρου 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 38, 9, δύο εποχές. Συγχαρητήρια. Και ευχαριστώ τους συναλλεύους που δούλεψαν για το θέμα αυτό με πολύ πίεση χρόνου. Ευχαριστώ για το έργο σας. Σημείο 5 καταπολέμηση της τρομοκρατίας και αντικατάσταση του, της, ε, του, της αποφάσεως πλαισίου του Συμβουλίου για καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Με εισηγείται την κυρία Χολμάγερ. Εγκρίνεται, θα εγκριθεί το σχέδιο γνωμοδότησης για, τις, και το, για το ξεκίνημα της, ε, των διοργανικών διαπραγματεύσεων και την ε, σύσταση της διαπραγματευτικής ομάδας. Υπάρχουν κάποια σχόλια, όχι. Υπάρχει και ένα επιπλέον σημείο. Οι συντηρητικοί σήμερα το πρωί ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία για το άρθρο 18. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 208 πρέπει να ζητηθεί η έγκριση από 15 μέλη, το ενεργών της Επιτροπής. Θέλω να, ελά... να ελέγξω αν υπάρχουν 15 συνάδελφοι που στηρίζουν το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας, αν θέλετε. Κρατήστε τα χέρια ψηλά. η τροπολογία 80 θα γίνει λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Άρθρο 1. Τροπολογία 205. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Δεκτή. Συμβαστική 11 ψηφοφορία. Ονομαστικά, ονομαστική ψηφοφορία που ζητήθηκε από το ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Όχι. Τώρα κλείνει. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Πάλι ονομαστικά μετά από έτοιμα του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 207 του απολογίας, παράγραφο 1, άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της Απορρίπτεται. Διακόσια τροπολογία στο άρθρο 2, άρχεται η ψηφοφορία. Διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 209, άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 209. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε τη 211 και τη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 210 το υπολογία ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το τοπολογία 212 για το πρώτο τμήμα. Γίνεται κατά τμήματα η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Πέρα ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα του 212. Άρχεται η ψηφοφορία. υπάρχει ένας σοσιαλιστής παραπάνω στην ψηφοφορία αυτή. Για οργανωθείτε. Okay, the vote is now closed and that is rejected. απορρίφθηκε για αυτό το τμήμα. Συνάδελφοι, προχωρούμε. 213. Τοπολογία άρχεται η ψηφοφορία. 213. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεκτή διορθώνει ο πρόεδρος. 214. Άρχεται η ψηφοφορία. Μόνικα. Μπορείς να βγάλεις το όνομά σου πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 205 το Ε, 215, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα έχουμε έναν παραπάνω στο ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 216. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 218, 219 και 222 που είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τρεις αυτές τροπολογίες. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτές. 223 τώρα. Ονομαστικά μετά από έτοιμα του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 224. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη Απορρίπτεται. 225. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Δεκτή. 226. Ψηφίζουμε. Πέρα τη Απορρίπτεται. 227. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 228 ονομαστικά μετά από αίτημα ΕΛΚ και Πρασίνων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 229. Ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Πάλι ονομαστικά μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2.30 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία Δεκτή. 231. Ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.32. Ονομαστική από το ΕΛΚ. Έναρξη. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 2-3-3 3 εναξη ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Ονομαστική κατά του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 234. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 239. Ονομαστική έτοιμα ΕΛΚΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 2.37, ονομαστική ε, των Πρασίνων. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε, διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 2.41, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία. 2.43 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚΑ. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Ονομαστική ζήτησε το ΕΛΚ. Χωριστή ψηφορία που ζήτησαν οι πράσινοι. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 261. Ψηφίζουμε. Α, έχουμε να ψηφίσουμε και το δεύτερο τμήμα, γιατί ήταν κατά τμήματα η προηγούμενη ψηφορία. Δεύτερο του, της συμβαστικής έξι ψηφίζουμε. Συγγνώμη, μας έχει, το Brexit μας έχει, μας έχει κάνει τα νεύρα πέρα της ψηφορίας. Εγκρίνεται. 2.61, έναρξη. Πέρας ψηφορία εγκρίνεται. 262. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 263 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 264 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 266 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 267 έναρξη. και πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. 268 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Κατά τμήματα οι πράσινοι το ζήτησαν και ονομαστική ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ε, το ΕΛΚ η πράσινη τη ζήτησε Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2, 8, 9. Ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απολύπτεται. 35 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Το έλκη και η πράσινη τη ζήτηση να ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τώρα τμήμα ψηφίζουμε. Πέρας. Ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 3, 0, 3 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Απορρίπτεται. 302. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκριέται. 305 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 307 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Σαράντα ένα. Ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.37 ψηφίζουμε. Πέρας. Τρία 3.40 ψηφίζουμε. Που είναι ίδια, ταυτόσιμη με την 44. Αν το ακούσετε συνάδελφοι, αν το δέχεστε αυτό, συνεχίζουμε κανονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 341 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. 342 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 343 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, όλες μαζί. Ψηφίζουμε. Πέρασε ψηφορίας. Απορρίπτεται. 3.49 ψηφίσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 3.50 ψηφίσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 3, 45 και 351 ταυτόσιμες, λέει ο πρόεδρος, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 352 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 353 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 354 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 355 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 356. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 357 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 358 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 359. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9. Ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚ. Ψηφίζουμε. Close. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 364. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 371 και 372. Η 371 είναι ονομαστική που αιτήθηκε το ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχετε ήδη ξεκινήσει. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 372. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 376. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 397. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 419 που είναι όμοια με το 413 και είναι ονομαστική ψηφοφορία. Τη ζήτησε το ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το τροπολογία 425. Unblock. 422, 23, 25, 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47. Είπε, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48. Είπε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 431 και 433 όμοιες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 432. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Η 432 καταπίπτει και πάμε στην 430. Ακυρώνεται το 432 και ψηφίζουμε για την 430. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 435-437 όμοιες. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 438 ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε το ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 56. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Βρισκόμαστε στις αιτιολογικές σκέψεις. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 ονομαστική που ζήτησε το ΕΛΚΑ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Άρχεται η ψηφοφορία. 69. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74 και 76 Ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 80 ονομαστική που ζήτησε το ECR. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Ονομαστική ψηφοφορία από το ΕΛΚ. Ζητήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 133. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 140. Συγγνώμη. Η 138, 140 και 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι ταυτόσημες. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 144. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται υπολογείο 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Δεκτή. Εκατόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 149 Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 200 τροπολογία. Και 151 ίδιες. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 153. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10. Ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα των Πρασίνων και του ΑΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 182 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 183. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 184. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 186. Άρχεται η ψηφοφορία. Διορθώνει ο 185. 185 τροπολογία ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 186. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Δεκτή. 197 όμοια με την 196-198. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 199. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Δεκτή. 201. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίες. Δεκτή. 27. Άρχεται ψηφοφορία. Διορθώνει ο πρόεδρος. 202 τροπολογία ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας δεκτή. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως το εποποιήθηκε. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. συνεχίζεται να είναι ανοιχτή. Ψηφίσατε όλοι οι συνάδελφοι. Μισό λεπτό. Θέλω να ελέξω αν η 219 τροπολογία έχει καταπέσει. 291, ε, συγγνώμη. Θέλω να μην τεθεί σε κίνδυνο το κείμενο. Θα ήθελα να ψηφίσουμε την τροπολογία 291 που δεν το κάναμε. Σε σελίδα 8. Δείτε τον κατάλογο ψηφοφορίας σας. 291. Δεν την ψηφίσαμε. Είναι ονομαστική η ψηφοφορία μετά από έτοιμα του ΕΛΚ που δεν ψηφίσαμε από ό,τι φαίνεται. Είναι, έχει ζητηθεί ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα δεν ψηφίσαμε, δεν έχει καταχωρηθεί. Παρακαλώ να γίνει ψηφοφορία για την 291 τώρα. Αν... Λοιπόν, συμφωνείτε όλοι ότι το ψηφίσαμε. Εντάξει. Ψηφίζουμε. Βρήκατε την σελίδα 8 που είναι η τοπολογία. Σελίδα 8. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη, δίκιο έχουν. Δεν μπορεί να ψηφιστεί. Ε, το, ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του κειμένου όπως το τοποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρα στις Δεν τελειώσαμε. Έχουμε κι άλλο. Εγκρίνεται το σχέδιο. 41 υπέρ 10, 4 κατά 10 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια πρέπει να αποφασίσουμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, την ε, εντολή και την διαπραγματευτική ομάδα. Αυτό απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία ε, βάσει του άρθρου 73. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένουμε μέχρι να γυρίσουν αυτοί που φεύγανε, να βάλουν την κάρτα τους ε, Ψηφίσατε. Εγκρίνεται. 47, 5, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και πάλι. Τώρα μπορείτε να φύγετε. Έχουμε κι άλλο ένα θέμα, συνάδελφοι. Θέλει να πει κάτι η συγγήτρια, συνάδελφοι. Μισό λεπτό. Να σας ευχαριστήσω όλους τους τους εισηγητές. Είχαμε μια πολύ καλή διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια ευχαριστεί τους ε, εμπλεκόμενους συναδέλφους ε, που ήταν σκιώδεις εισηγητές. Uh, Συνάδελφοι, έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αν θέλετε να φύγετε, παρακαλώ να το κάνετε ήσυχα. Um, can we move Συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 6 παρακαλώ. Colleagues, um, we moved to... Συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 6, που είναι οι, τρεις, οι τρίτες χώρες, των οποίων οι πίκοοι πρέπει να διαθέτουν θεώρηση για την διέλευση από τα εξωτερικά σύνορα και αυτές οι χώρες τις οποίες δεν απαιτείται μια τέτοια θεώρηση. Εξετάζουμε την, το σχέδιο έκθεσης. Η, η Μαρία Γκάμπριελ είναι η συγγήτρια. Ζητώ συγγνώμη για τον ε, θόρυβο και ζητώ συγγνώμη που έπρεπε να συζητήσουμε το θέμα τόσο αργά. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι μία νομοθετική πρόταση για να τροποποιήσουμε τον κανονισμό 539 του 2001 που μεταφέρει την ε, Γεωργία στην ε, κατάσταση με τις χώρες που δεν απαιτούν θεώρηση ότι η άρση της θεώρησης γίνεται λόγω της ε, ύπαρξης βιομετρικών διαβατηρίων. Εντάξει, λίγο θόρυβο συνάδελφοι να τον κάνετε, αλλά όχι να συζητάτε παράλληλα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της άρσης της υποχρέωσης θεώρησης. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Στις ε, 25 Απριλίου του περασμένου έτους, η, το, που μόλις μας πέρασε η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της στην Επιτροπή με παρουσία των εκπροσώπων της Γεωργίας που συμμετείχαν στη δεύτερη συνάντηση της ε, Επιτροπής ε, της Κοινοβουλευτικής Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία. Η πρόταση έρχεται μετά από μια, ε, έναν διάλογο που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012. Η Κομισιόν παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης για την Απελευθέρωση από την υποχρέωση για τη βίζα. Έχουμε την τέταρτη και τελευταία έκθεση προόδου. Φαίνεται από αυτήν ότι έχει υπάρξει απαραίτητη πρόοδος και σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία παρουσίασε η Κομισιόν την πρότασή της. Ε, αυτό έχει φυσικά επιπτώσεις και σε άλλα θέματα αντίστοιχα για θεωρήσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στην κυρία Γκάμπριελ που ήταν η για αυτό το θέμα της Γεωργίας και μετά στους Σκιώδης και όποιο άλλο μέλος θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Γκάμπριελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χαρά μου σήμερα που σας παρουσιάζω το σχέδιο έκθεσης για την απελευθέρωση του καθεστώτας θεώρησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να επανέλθω στο πλαίσιο της πρότασης ως έχει. Καταρχάς, ο διάλογος για την απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρησης ε, ε, και το καθεστώς ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Γεωργίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012. Υπήρχε μια ε, μικρή διάρκεια τέτοια ε, αναμονή για να βγουν τα βιομετρικά διαβατήρια. Πρόκειται λοιπόν να απελευθερέσουμε την μόνο για τους υπηκόους που έχουν βιομετρικό διαβατήριο την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ του 2013 και της 18 Δεκεμβρίου του 2015 είχαμε τέσσερις εκθέσεις ε, εκ των οποίων προέκυψε αυτή η πρόταση. Άρα η Γεωργία όχι μόνο εκπλήρωσε όλα τα κριτήρια, αλλά και οι αρχές της Γεωργίας πήγαν ακόμα παραπέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις με νέες ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες από τότε που Ξέδωσε η Κομισιόν την τελευταία της έκθεση. Έκαναν λοιπόν όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες και γι' αυτό πρέπει να τους συγχαρούμε και να στείλουμε αυτό το θετικό μήνυμα για τις προσπάθειες των αρχών. Επίσης, ε, η απελευθέρωση από την υποχρέωση τη θεώρησης είναι μεταξύ, ένα άλλο βήμα στην προσπάθεια προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργίας που θα ωφελήσει του πολίτε και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργία. Η Γεωργία είναι ένα στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία και τη Ανατολική Εταιρική σχέση πιο συγκεκριμένα. Σήμερα, μεταξύ άλλων, έχουμε και αυτή την συνάντηση την 4η Ιουλίου, ε, κατά την οποία μπορούμε να υπογράψουμε να υπογραμμίσουμε ότι την 1η Ιουλίου που ξεκίνησε η Συμφωνία Σύνθεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε ε, όλα τα βήματα έτσι ώστε να υπογραμμισουμε οτι την 1 η ιουλιου που ξεκινησε η συμφωνια συντασης μεταξυ ευρωπαικης ενωσης και γεωργιας μπορεσαμε να ολοκληρωσουμε ολα τα βηματα ετσι ωστε να εχουμε μια συμφωνία που θα είναι και αυτή κομμάτι της γενικότερης προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία που θα προσπαθήσουν μαζί να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να έχουμε και πολιτική και οικονομική προσέγγιση. Η εξαίρεση από την υποχρέωση για τη θεώρηση πρώτα απ' όλα ωφελεί τους πολίτες. Δεν πρέπει ποτέ να χάνουμε από τα μάτια μας τους πολίτες. Οι Ευρωπαίοι, οι πολίτες μπορούν να μπουν στη Γεωργία χωρίς βίζα. Σήμερα λοιπόν ε, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα πρέπει να επιτρέψουμε την απελευθέρωση από τη θεώρηση και την προσέγγιση και εμβάθυνση των κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ ε, των δύο μερών. Πρόκειται για κάτι που περιμένουν από εμά ένα συγκεκριμένο μέτρο για την εντατικοποίηση των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων αλλά και του πολιτικού διαλόγου που περιλαμβάνει και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα κριτήρια που μας επέτρεψαν να κάνουμε αυτή την πρόταση είναι κριτήρια που έγιναν σεβαστά. Είπα ότι οι αρχέ πήγαν πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσει και εμείς ως κοινοβούλιο συνεχίζουμε να εκφράζουμε την άποψή μας ότι πρέπει να ενισχυθεί ο διάλογος, να συνεχίσει και να δούμε τι θα γίνει μετά από αυτό. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τις βασικές μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί σήμερα έχουμε ένα σχέδιο δράσης το οποίο μας επέτρεψε να εξετάσουμε τη θεσμική και πολιτική κατάσταση και να πούμε ότι είναι σχετικά σταθερή. Όμως το σχέδιο δράσης αποδείχθηκε και ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόθεση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων μεγάλης κλίμακα, ιδιαίτερα στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Λοιπόν, ε, θα μας βοηθήσει τώρα να ε, έχουμε πιο ανοιχτέ σχέσεις, να μιλάμε καλύτερα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γεωργία μέσα στα πλαίσια του ετήσιου διαλόγου που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτά τα πλαίσια να επανέλθω σε κάποια νούμερα που ήταν αντικείμενο συζήτησης όσο ε, προετοίμαζα την έκθεσή μου. Ξέρουμε ε, πόσο μας ενδιαφέρει η κινητικότητα και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν σε επίπεδο μετανάστευσης και ασφάλειας. Παρόλο που υπήρχε μια αύξηση των ετοιμάτων, όμως παρέμεινε σταθερός ο αριθμός της απόρριψης το 2015. Το 2014, σύμφωνα με τη Eurostat, ε, μειώθηκε κατά 61% σε σχέση με το 2013 και 50 περίπου σε σχέση με το 2015 ο αριθμός των ανθρώπων που πέρασαν τα σύνορα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα ανάλυσης ε, που θα μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την μετανάστευση συνολικά, να βρούμε τους κινδύνους, να δούμε σε τι βαθμό ε, επιτυγχάνουμε αυτά που ε, πολλοί μας ενδιαφέρουν. Οι αρχές της γεωργίας λοιπόν ε, έχουν όπως είπα θέσει σε εφαρμογή πολλά εργαλεία που μας επιτρέπουν να έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για τους ε, πολίτες, ε, για τα δικαιώματά τους και για τις υποχρεώσεις διάπασης χωρίς βίζα των συνόρων. Να ευχαριστήσω λοιπόν ε, και να πω ότι σήμερα υπάρχει και μια συμφωνία με τη Europol. Πρέπει να συγχαρούμε τη Γεωργία γι' αυτό, γιατί μπόρεσε να συμβάλλει επικοδομητικά στον αγώνα κατά της ε, του οργανωμένου εγκλήματος. Τέλος, να επιμείνω σε κάτι που συστήνω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΑ είναι ε, να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής, διότι εξ αρχής θεωρώ ήμασταν πολύ ξεκάθαροι στη μέθοδο που ακολουθήσαμε. Είπαμε ότι μόλις εκπληρωθούν τα κριτήρια σε ατομικό επίπεδο με βάση ε, τις προσπάθειες που έκανε η Γεωργία, θα πούμε ε, ότι εγκρίνουμε, παρόλο που φυσικά υπάρχει μια διαδικασία που συνεχίζει και υπάρχουν και εργαλεία που θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Τελειώνω λέγοντας ότι αυτό που γίνεται στη Γεωργία έχει μεγάλη σημασία για εμάς, η ασφάλεια, η σταθερότητα. Η ευημερία αυτή τη χώρας επηρεάζει όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουμε κοινό συμφέρον να συνεργαστούμε στενά και να υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό μέσο την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Γεωργία. Σήμερα λοιπόν στέλνουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα στους πολίτες της Γεωργίας για να μπορέσουν να συνεχίσουν με την πεποίθηση που μας έδειξαν ε, ότι έχουν να ακολουθήσουν το σωστό δρόμο ε, την ε, πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Γκάμπριελ. Τώρα έχουμε μια σειρά σκιωδών και άλλους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Παρακαλώ να μιλήσετε με τη σειρά ε, που ε, έγινε η αίτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Μαρία. Θέλω πολύ σημαντικό την διαδικασία ελευθέρωσης των θεωρήσεων να την κρατήσουμε ζωντανή και αξιόπιστη. Όπως είπατε, πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική και πολιτική συνεργασία, τις επαφές μεταξύ των λαών και συναφώς υποστηρίζω την αποψή σας. Συγχαίρω επίσης τις αρχές της Γεωργίας για τις προσπάθειές τους. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την πρόοδο όταν είναι πρόοδος και όταν υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσει και τα κριτήρια. Είχα ασχοληθεί με το θέμα και στα Δυτικά Βαλκάνια και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ο κόσμος καταλαβαίνει. Δηλαδή κάθε χώρα έχει τα δικά της φυσικά πλέον πλεονεκτήματα. Όταν πάρω κάποιο σημειώνει πρόοδο και πλήρει τα κριτήρια να το αναγνωρίζουμε. Και αυτό θα κάνει την πολιτική μας για τις θεωρήσεις διατηρήσιμη, βιώσιμη. Την περασμένη φορά μιλήσαμε και για το Κοσμοπέδιο, για την Ουκρανία, μετά την Τουρκία. Εδώ δεν πρόκειται για πολιτικό ζήτημα. Κρίνουμε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια, πολύ απλά. Έτσι, συμφωνώ και υποστηρίζω ολόθερμα την επέκταση του καθεστώτος ε, στην Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και εγώ να δηλώσω την υποστήριξη της πολιτικής μας ε, ομάδας υπέρ της ε, έκθεσης η οποία συνηγορεί υπέρ της ελευθερίας του καθεστώτος τη Γεωργία με επικεφαλής Μαρία σύμφωνα με τους προλελήσαντες πρώτον η Γεωργία ικανοποίησε όλες τις απαιτήσεις πλήρει όλα τα κριτήρια σημείωσε την απαιτούμενη πρόοδο και μπορεί να απολάβει της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων. Είναι λογικό λοιπόν, πολιτικός και άλλος, να συνεχίσει τη διαδικασία. Εν παρόδο, να χαιρετήσω την καλή θέληση που επικράτησε από όλε και προς όλες τις κατευθύνσεις και δύο από τις αρχές της Γεωργίας. Η Γεωργιανή ήταν πολύ πρόθυμοι προχώρησαν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες υπερβαίνουν μάλιστα και τις προσδοκίες μας. Όπως είπε και η Μαρία Γκάμπριελ πριν από λίγο, πρόκειται για μια διαδικασία, όντως. Η πολιτική μου ομάδα πιστεύει ότι οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν δείχνουν ότι γίνεται προσπάθεια ότι η χώρα εξελίσσεται πρέπει να φροντίσουμε αυτά να συνεχιστούν και μάλιστα να παγιωθούν και μιλώ για θέματα όπως η προσφυγή στην δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ο τύπος και το καθεξής. Όπως είπαν και οι για άλλη μια φορά, η Γεωργία βεβαίω είναι σύμμαχος στρατηγικός, αλλά η επέκταση αυτή, η ελευθέρωση των θεωρήσεων είναι θέμα σημαντικό για τους πολίτες της Γεωργίας. Κρατώ όμω τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέση μας με την Γεωργία στο πλαίσιο της Ανατολική Γειτονία. Να μαθαίνουμε λοιπόν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της Ένωσης και του Νοτιού Καυκάσου. Είναι το οποίο είναι σημαντικό για αυτές τις χώρες, αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικό, για μας. Γι' αυτό λοιπόν και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζουμε 100% την εν λόγω έκθεση. Ευχαριστώ. Βαλέρο. Νομίζω ότι με κάλυψαν οι προηγούμενοι. Χαίρομαι που οι Γεωργιανοί θα ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση. Και για μένα μάλιστα είναι πολύ θετικό το ότι μπορούμε να πηγαίνουμε στη Γεωργία χωρίς θεώρηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση. Οι ανησυχίες που αισθάνθηκα κατά τη διάρκεια της συζήτησης έχουν σχέση με εξελίξεις οι οποίες είναι εικασίε περί μελλοντικών εξελίξεων που θα δούμε αν θα συμβούν, οπότε ε, είμαι θα υπέρ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ την Μαρία Γκάμπριελ ως ε, εισηγήτρια αλλά και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Εξαιρετική η έκθεση. Καλώς δίνουμε ένα θετικό σήμα, ένα θετικό μήνυμα προς τους Γεωργιανούς που περίμεναν την ελευθέρωση, διότι οι Γεωργιανές αρχές εκπλήρωσαν όλα τα κριτήρια μετά και από την συμφωνία με την Γεωροπόλη. Στην Γεωργία θα γίνουν συντομαστητά τα πλέον εκτίματα από την ελευθέρωση του καθεστώτος. Υποστηρίζω λοιπόν την εξέλιξη αυτή ε, Νομίζω δουλέψαμε πολύ γρήγορα και ικανοποιητικά. Και η Μαρή Κριστίν Βεργιά. Μαρή Κριστίν. Πολύ σύντομα καλύφθηκα ήδη από τους προλαλήσεντες και εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων εκ μέρους και της ομάδας μου που είναι η υπέρ της ελευθέρωσης των θεωρήσεων, ιδιαίτερα με τις χώρες της γειτονίας και δι, εφόσον, όταν και εφόσον οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαύουν το ίδιο προνόμιο. Πρόκειται για αμοιβαιότητα που μου φαίνεται απολύτως φυσικό. Έχουμε μετά και την Τουρκία, μην ξεχνάτε. Οπότε εγώ προκειμένου εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρώτη που σημείωσε η Γεωργία όσον αφορά το δικαίωμα στη χορήγηση ασύλου και όσον αφορά το θέμα της ηθαγένειας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ που παραμείνατε ως αυτήν την ώρα για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Κύριε Γκάμπριελ, μια κατακλίδα, όχι. Πολύ ωραία προθεσμία. 14 Ιουλίου 12 το μεσημέρι για την κατάθεση τροπολογιών. Θέλετε να πείτε ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ λέει, κύριε Καμπρίλ. Ευχαριστώ στους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ και όσους έλαβαν τον λόγο. Σε ευχαριστώ το μήνυμα που στέλνουμε. Είναι κάτι το οποίο δίνει σαφές μήνυμα στις χώρες της γειτονίας. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Στα διάφορα κάτι άλλο όχι. τη συνάδελφοι, θα πούμε 7 Ιουλίου, 11 Ιουλίου, 12 Ιουλίου, Στρασβούργο, Βρυξέλλες και Βρυξέλλες αντιστοίχως. Συνεχίζουμε με την συνάντηση των συντονιστών. Παρακαλώ όσοι δεν έχουν δουλειά να αναχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ.